Dear Αγαπητοί συνάδελφοι, ας ε, ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας ε, με την έγκριση της αμυρίσιας διάταξης. Όπως ξέρετε, αυτό το πρώτο σκέλος της συνάντησής μας είναι κοινή επιτροπή με την Επιτροπή Προϋπολογισμών. έγκριση λοιπόν της ε, ημερήσιας διάταξης και θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Περβάνσο Περές, ε, είναι η νέα συντονίστρια των ε, Σοσιαλδημοκρατών. Πάμε τώρα στις ανακοινώσεις του Πρόεδρου που δεν υπάρχουν ανακοινώσεις Πρόεδρου. Κατόπιν τούτου ε, πάμε στην έγκριση των πρακτικών της 13 ε, ε, Τρίτης, τέλος πάντων των πρακτικών του Απριλίου. Και προχωράμε στην εξέταση του σχεδίου έκθεσης του κυρίου Μπέγκε και της Περβάνς Μπερές για τις ε, δημοσιονομικές ε, δυνατότητες για την Ευρωζώνη. Όπως ξέρετε, ε, οι συγητές υποβάλλουν ενδιαφέρουσα και φιλόδοξη έκθεση, σχέδιο έκθεση. Είχαν επίσης ένα γύρο σημαντικών αποστολών σε κάποιες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες καθώς επίσης και κάποιες σημαντικές συνεδριάσεις με την πιο πρόσφατη, με τον κύριο Ρέγκλινγκ. Πολλή δουλειά έχει γίνει λοιπόν ήδη, πολλή προετοιμασία και θα ήθελα να σας συγχαρώ και να σας ευχαριστήσω. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα. Ε, έχουμε πολύ ε, σημαντικό προπολογισμό, προπολογισμό για την ενιαία αγορά αλλά και για το ενιαίο νόμισμα. Οπότε mm. είναι ακριβώς αυτό το ζήτημα. Πώς μπορούμε να λάβουμε υπόψη όχι μόνο την ενιαία αγορά αλλά και το ενιαίο νόμισμα και πώς μπορούμε να συμπληρώσουμε τον προϋπολογισμό της ενιαίας αγοράς με το προϋπολογισμό για το ενιαίο νόμισμα. Θα ήθελα να δώσω το λόγο λοιπόν στην εισηγήτρια Περβάνος Μπερέζα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Στο πλαίσιο του άρθρου 55 και τη κοινή συνεργασίας ανάμεσα στις δύο επιτροπές μας είναι μια σημαντική φάση όπου μετά από την παρουσίαση δύο εγγράφων εργασίας τα οποία είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε στην προηγούμενη συνεδρίαση σήμερα σας υποβάλλουμε το σχέδιο έκθεσης το ίδιο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 Le point de départ, euh, vous l'avez... Κοινή προσέγγιση. Ε, στην πράξη, κύριε Πρόεδρε, σήμερα ε, βρισκόμαστε ενώπιον ε, μιας προφανούς κατάστασης, ότι δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ποτέ δεν ξαναεξέτασε την κατάσταση μετά από την αλλαγή προς το ευρώ. Όμως το πέρασμα στο ευρώ είχε επιρροή τόσο στις επενδύσεις όσο και στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Και αυτό δεν απετέλεσε ποτέ αντικείμενο μελέτης αντικτύπου. Η ίδια η κρίση όμως έδειξε πόσο ευάλωτη είναι η κατάσταση για το ευρώ. Γι' αυτό και εμείς οι συνεισηγητές είμαστε απόλυτα πεπισμένοι ότι όταν μιλάμε για την ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, ένας από τους πυλώνες αυτής της ολοκλήρωσης είναι η δημιουργία ενός δημοσιονομικού ε, μέσου συγκεκριμένου με ε, κονδύλια για την Ευρωζώνη, όπως ε, ε, είχε προτείνει το Κοινοβούλιο μας από το 1998 σε ένα ψήφισμα του, το οποίο πρότεινε η Επιτροπή αυτή, η Οικονομική και Νομισματική Επιτροπή, υπό την ευθύνη του συναδέλφου Μέτεν, που δείκνει ότι για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε ασυμμετρικά σοκ, ε, το ευρώ θα έπρεπε να έχει ένα ταμείο σταθεροποίησης, έλεγε από τότε. Οι συγκητές σας είναι επίσης πεπισμένοι γι' αυτό, ότι υπάρχουν δηλαδή χρήσιμα στοιχεία στην έκθεση των πέντε Προέδρων. Απλά είμαστε επίσης πεπισμένοι ότι η δεύτερη φάση, που είναι η φάση που μας απασχολεί σε αυτή τη συζήτηση, δεν μπορεί να ε, την αναμένουμε με σταυρωμένα χέρια ότι θα πρέπει να προετοιμάσουμε αυτή τη δεύτερη φάση των πέντε Προέδρων γιατί και η ίδια η έκθεση των πέντε Προέδρων χρειάζεται κάπου και, που και που να συμπληρωθεί με βάση τις εργασίες που γίνονται έκτοτε. Δεν θέλω να μακρηγορήσω στην ε, αρχική μου εισήγηση γιατί θα ήθελα ε, να έχουμε μια πλούσια ανταλλαγή απόψεων και ξέρω ότι είναι ένα θέμα το οποίο είναι ιδιαίτερα αγαπητό στους συνάδελφους αλλά θα ήθελα να σας παρουσιάσω τη γενική προσέγγιση ε, που, μας, που προτείνουμε. Ξεκινώντας λοιπόν από αυτή την έλλειψη της λειτουργίας, τα προβλήματα λειτουργίας της Ευρωζώνης, θυμήσαμε επίσης ότι το Κοινοβούλιο από το από, ε, μάλλον ανέκαθεν ζητά να, να ενσωματωθεί ο μηχανισμός σταθερότητας στη κοινοτική μέθοδο όπως την αποκαλούμε και παρατηρούμε ότι πέρα από τα όσα εμεί θελήσαμε αυτό εγγράφεται και στη δεύτερη φάση όπως την περιγράφει η έκθεση των πέντε προέδρων. Εκινώντας από αυτό, θεωρούμε ότι ο τρόπος με τον οποίο ο μηχανισμός σταθερότητας θα ενσωματωθεί στην κοινωτική μέθοδο και θα διαρθρωθεί όχι μόνο με τον προπολογισμό της Ένωσης αλλά και με το πολιετές ε, ε, δημοσιονομικό πλαίσιο. Χρειάζεται λοιπόν αυτό όλο να τελειοποιηθεί και από αυτό έχουμε διάφορες προτάσεις. Με πρώτη ότι αυτό θα πρέπει να γίνει πέρα από το πλαίσιο και το κατόφλι που προβλέπεται από το PDP. Έχουμε τρεις λειτουργίες που πιστεύουμε ότι πρέπει να καλύπτονται από αυτές τις δημοσιονομικές δυνατότητες της Ευρωζώνης. Ο πρώτο είναι η σύγκληση, το δεύτερο είναι η απορρόφηση των ασυμμετρικών σοκ και το τρίτο είναι η δυνατότητα να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε συμμετρικά σοκ. Κατά την ανάγνωση της έκθεσης και μετά από την ε, ε, συσσόρευση αποδείξεων μέσω διαφόρων ανταλλαγών απόψεων κατά τη διάρκεια της σύνταξης έκθεσης, θεωρούμε ότι αυτές οι τρεις λειτουργίες θα έπρεπε να καλύπτονται από δημοσιονομικά και οικονομικά μέσα σε παραπληρωματικά. Αυτό σημαίνει ότι ε, για τον πρώτο στόχο, τη σύγκληση, που είναι απαραίτητη για να εξασφαλιστεί η στάθεια της Ευρωζώνης σε διάρκεια, αλλά και έτσι ώστε οι δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις στην Ευρωζώνη να μην υποτιμούνται διαρκώς όπως σήμερα, πιστεύουμε ότι πρέπει να βρούμε μέσα στον προπολογισμό της Ευρωζώνης και με την ευκαιρία της αναδιατύπωσης του PDP εργαλεία τα οποία θα επιτρέπουν να βελτιώνεται η σύγκληση. Και γι' αυτό το λόγο, πέρα από το οικονομικό εργαλείο το ίδιο, ε, προτείνουμε να ξανάρθουμε σε μια ιδέα που εσείς ο ίδιος, κύριε Πρόεδρε, μαζί με τον Έλμαρ Μπρόκ και τον Κίφερ Χόφστατ είχατε υποβάλει στην προηγούμενη εντολία ως συμβολή των ΣΕΡΠΑ στην σύνταξη της έκθεσης των τεσσάρων Προέδρων, να βρούμε δηλαδή έναν κώδικα σύγκλησης που βασιζόταν τα κριτήρια του Μάστριχτ που είχαν οδηγήσει σε μεταρρυθμίσεις πολύ ουσιαστικές στα κράτη-μέλη καθώς και μια σημαντική ε, ε, ε, ιδιοποίηση από πλευρά των κρατών μελών της μεταρρύθμισης αυτής. Ε, αντί να έχουμε δηλαδή κυρώσεις ή ποινές, ε, ήταν πιο αποτελεσματικό αυτό παρά οι μηχανισμοί που τελικά θεσπίσαμε μετά από την μετάβαση στο ευρώ. Η δεύτερη λειτουργία της αντιμετώπισης απορρόφησης των ασυμμετρικών ε, σοκ από την άποψη των πυρογνωμόνων, των οικονομολόγων είναι ίσως η πιο σημαντική λειτουργία, η καρδιά της συζήτησης. Αλλά το βάζουμε θελημένα ως δεύτερο στόχο και εδώ τίθεται το θέμα της διατήρησης της δραστηριότητας του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, αλλά μια κοινοτική προσέγγιση. Και αυτός ο μηχανισμός να συμπληρωθεί, που, αυτός ο μηχανισμός που για την ώρα είναι ένας μηχανισμός ε, περιλαμβάνει όρους και ορίζει αναπερίπτωση να συμπληρωθεί από μια αυτόματη προσέγγιση, πράγμα που επιτρέπει να περιοριστούν τα στοιχεία συζήτησης ή αμφισβήτησης σε φάσεις έντασης και δίνει τη δυνατότητα στους φορείς να αποκαταστήσουν τη λειτουργία της ζώνης. Και οι δυο μηχανισμοί που συζητώνται εδώ και πολλά χρόνια και τους οποίους ε, παραθέτουμε είναι αυτό που λέμε το Ταμείο για τις ε, δύσκολες μέρες, δεν ξέρω ακριβώς πώς το λέμε στα γαλλικά, αλλά Rainy Day Fund το Ταμείο για τις δύσκολες μέρες και εκείνο το Ταμείο για τη μήνυμο με επίδομα ανεργίας. Τρίτη ε, λειτουργία, η απορρόφηση συμμετρικών σόκων, που πιστεύουμε ότι το υφιστάμενο διατακτικό θα πρέπει να συμπληρωθεί. Δηλαδή, εφόσον θα συμφωνήσουμε για αυτέ τι τρει λειτουργίε και το μηχανισμό χρηματοδότηση αυτών των τριών λειτουργιών, θα πρέπει να εμβαθύνουμε και στο θέμα τη διακυβέρνηση. Και εδώ έχουμε ένα σωρό προτάσει, επί των οποίων είμαι βεβαία ότι οι συνάδελφοι θα σχολιάσουν και θα συμβάλλουν στον κοινό μας προβληματισμό. Σας ευχαριστώ πολύ για την ε, εισήγηση αυτή. Και τώρα περιμένουμε τον κύριο Μπέγκε, εξ ονόματος του ΕΛΚΑ, αλλά μεταξύ θα δώσω το λόγο στον κύριο Μπάλτς. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Μου ζήτησε ο σκιώδης μας να πάρω εγώ το λόγο γιατί έπρεπε να γιορτάσετε την 40η επέτειο της ρίσης του κόμματός μας ε, στο Λουξεμβούργο, καθότι είναι ο εκπρόσωπος της ομάδας. Είναι λοιπόν στο Λουξεμβούργο και γι' αυτό μου ζήτησε να πάρω το λόγο στη θέση του και φυσικά δεν έχω κανένα πρόβλημα να τον αντικαταστήσω. Μου είπε λοιπόν ε, ότι είχε κάποιες ανησυχίες ε, αφού διάβασε την έκθεση για την ε, δημοσιονομική ικανότητα, διότι θεωρεί ότι η έκθεση αυτή υπονομεύει ορισμένα στοιχεία του νομικού πλαισίου της Ένωσης και πολλές φορές ε, είναι και παραπλανητική, σε ό,τι αφορά ιδίως τα εξή σημεία. Πρώτον, δεν ορίζει σαφώς ή ορθώς την ΟΝΕ. Δεύτερον, θεωρεί ότι ο ΝΕ ναι και το ευρώ είναι, η κρίση, ε, είναι υπεύθυνοι για την κρίση του δημοσίου χρέους και όχι οικονομική κακοδιαχείριση κάποιων κρατών χωρών. Ε, υπήρξε βέβαια και αυτό. Ε, κάποιες χώρες δεν εφάρμοσαν τις ε, μεταρρυθμίσεις, άλλοι αύξησαν τις δημόσιες δαπάνες ε, χωρίς να αυξήσουν και την παραγωγικότητα. Υπήρξαν και κάποια πολύ υψηλά επίπεδα δημοσίου χρέου και μακροοικονομικέ ανισορροπίε που σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για δεκαετίες δεν άφησαν περιθώρια λιγμών σε αυτές τις χώρες όταν έπληξε, όταν χτύπησε η κρίση. Ναι, μάλλον ήταν μεγάλη αυτή η πρόταση που σας διάβασα. Ο Ζίγκφριτ όμως έτσι τα έγραψε, τι να κάνουμε. Κατά την άποψη του Ζίγκφριτ δεν ε, παρουσιάζεται παρκώς η κατάσταση για την κρίση. Under the current treaty framework. Έχουμε ένα μέσο, case. Έχουμε τα άρθρο 195 της ε, ε, τη ρήτρα για το known bailout όπως λέγεται, που απονομεύεται. Το δικαστήριο λέει ότι δεν μπορεί η Ένωση να αναλάβει τα θεσμικά τη όργανα νέα καθήκοντα, νέε αρμοδιότητε. Γι' αυτό απαιτείται αλλαγή των συνθήκων. Επίση, δεν αναφέρεται στην έκθεση το γεγονό ότι η δημοσιονομική ικανότητα θα είναι περιορισμένη και δεν θα μπορέσει να σταθεροποιήσει τα μεγάλα κράτη-μέλη της Δεν θα πρέπει στόχο τη δημοσιονομική ικανότητα να είναι να σώζει χώρε που βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση γιατί υπάρχει ο ESM, ο Μηχανισμός ε, Μουσικής Σταθερότητας. Και υπάρχει και το άρθρο 125, συγγνώμη, άρθρο για το non-bailout. Αλλά δεν αναφέρεται αυτό το άρθρο στην έκθεση. Επίσης αναφέρεται μετάβαση από το ESM σε ένα Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο που θα το διαχειρίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά αυτό δεν είναι δυνατό με βάση το εφιστάμενο νομικό πλαίσιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Απαιτείται και γι' αυτό αλλαγή τη συνθήκη. Η έκθεση προτείνει επίση τη δημιουργία, ε, την, ε, τον ορισμό μάλλον ενό Υπουργού Οικονομικών. Αλλά λέει ότι θα πρέπει να είναι αρμόδιο για τα οικονομικά, αλλά και θα είναι και πρόεδρος του Eurogroup. Εμείς αυτό πρέπει να το απορρίψουμε. Αυτή είναι η άποψη του Ζίγκφριτ. Επόμενο Μετά την παράγραφη 23, fiscal capacity αντικαθίσταται από το ESM EMF. E Πάλι αυτό όμως μπορεί να γίνει μόνο με αλλαγή της συνθήκης. Η δημοσιονομική κάνοτητα δεν μπορεί να επιτελέσει τη λειτουργία το ESM. Το λέει ξεκάθαρα και στον πέντε πρόεδρων. Το να γίνει σε ESM, EMF, δημοσιονομική ικανότητα, όπως αναφέρεται στην έκθεση, υπονομεύει τη λειτουργία αυτού του μέσου και δεν θα μπορεί να προωθήσει τις ερωτικές μεταρρυθμίσεις, όπως προτείνει στον πυλώνα 1. Επόμενο σημείο. Τρεις πυλώνες προτείνονται στην έκθεση. Μόνο πυλώνας 1 δηλαδή να δοθούν κίνητρα για διαφορετικέ μεταρρυθμίσεις. Αυτό μόνο μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς αλλαγή των συνθήκων. Είναι περιορισμό και το μέγεθο. Άρα δεν μπορεί να απορροφήσει ασυμμετρικά και συμμετρικά σοκ και να σταθεροποιήσει την Ευρωζώνη συνολικά. Και πού μπορεί να εφαρμοστεί, σε πόσε περιπτώσει ταυτόχρονα. Επίση θα έλεγε ο κύριο Ζίγκφριντ Μόζον ότι θα πρέπει να εστιάσουμε σε στόχου που μπορούμε να πετύχουμε. Τελευταίο του σχολείο είναι ότι ο πυλώνα 2 είναι μια απλή προθέσεων. Δεν περιγράφει. Τι είναι αυτό το ταμείο για δύσκολους καιρούς, αυτό το Rainy Day Fund και αυτό το πρόγραμμα για το ευρωπαϊκό επίδομα δεν αναφέρεται λεπτομέρειε. Πώ μπορούν να αποφευθούν οι ηθικοί κίνδυνοι. Δεν αναφέρεται κάτι σχετικό. Και επειδή υπάρχουν αυτέ οι ασάφειε και ε, όλα αυτά τα προβλήματα, δεν είναι δυνατόν να το αποδεχθούμε αυτό. Άρα η μόνη λύση που δίνει η έκθεση στα τρέχοντα οικονομικά προβλήματα τη Ευρωζώνης είναι η δημιουργία μιας ένωσης μεταφορών πιστώσεων και αυτό το ταμείο ε, για τις δύσκολες μέρες ή το, το επίδομα ενεργείας. Δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστεί κάτι τέτοιο όμως, αν δεν αλλάξει η συνθήκη και αντιβαίνει εντελώ οποιαδήποτε τέτοια πρόταση με τη θέση της πολιτικής μας ομάδας. Αυτά ήθελε να πει ο Ζίγκριτ Μόζαν, αυτά μου έδωσε τουλάχιστον να σας διαβάσω. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Για το νομικό σκέλος Έχω κάποιες παρατηρήσεις για αυτά που λέει ο κύριος Μουρισάν, αλλά να δώσω καταρχάς τον συνεισηγητή κύριο Μπέγκε και να τον καλωσορίσω. Uh, my Eurostar had a huge delay which was not planned. Uh, I just uh, took note of the last uh, remarks from Mr. Mr. from Siegfried Muresan. Uh, to make it very clear,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 άλλη γλώσσα βγαίνει τα ελληνικά. Ε, κοιτάξτε, η γυναίκα μου που είναι Ελληνίδα μου λέει ότι ε, Είναι λοιπόν σημαντικό ε, να δώσουμε κάποια επαγγελματική μορφή σε όλα αυτά τα εργαλεία είναι λοιπόν ένας, ένα ενδιαφέρον θέμα και πρέπει να δούμε κατά πόσον όλα αυτά μπορούν να διευρυνθούν στο πλαίσιο του επόμενου EFF. Εγώ θα ήθελα απλά να σας πω ότι το ε, νομικό πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων ήδη προσφέρει κάποιες δυνατότητες τουλάχιστον όσον αφορά στην εφαρμογή και στην ε, αντίδραση ε, ορισμένων, σε ορισμένες καταστάσεις. Όλα αυτά τα χρησιμοποιούμε παρκώς, ναι ή όχι. Και πάλι, για να είμαι απόλυτα σαφές, τουλάχιστον όσον αφορά στο ρόλο της δημοσιονομικής ικανότητας. Όσο λιγότερο κεφαλαϊκή ένωση και τραπεζική ένωση υπάρχει ή δεν υπάρχει, τόσο περισσότερο χρειαζόμαστε μία ε, δημοσιονομική ικανότητα. Και αυτή, η σχέση, αυτή τη σχέση δεν μπορούμε να την αγνοήσουμε. Ε, νομίζω το Κοινοβούλιο ε, είναι δεσμευμένο και στους τέσσερις πυλώνες που ανέφεραν οι πρόεδροι. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία από αυτού. Το δεύτερο, όσον αφορά το ESM, η μετατροπή του σε Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο με τη δυνατότητα λήψης αποφάσεων και ισχυρή διακυβέρνηση, επ' αυτού, κατά την άποψή μου, πρέπει να είναι απόλυτα σαφές ότι αυτός, αυτό το προσετευτικό τείχος ε, που υπάρχει δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Σε αυτό το πλαίσιο μιλάμε για την ε, δημοσιονομική ικανότητα συμπεριλαμβανομένου και του νομισματικού ταμείου. Μιλάμε για μια δημοσιονομική ικανότητα η οποία ε, μπορεί να επιληφθεί όλων αυτών των συμπληρωματικών προγραμμάτων, βέβαια με όρους ε, για τα κράτη-μέλη, για να αποφεύγονται ε, τα σοκ. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι κατά πόσον η διαχείριση ενός τέτοιου ταμείου ε, μπορεί να γίνει από το EFM ή από το νομισματικό ταμείο. Πρέπει όμως να υπάρχει σαφής διαχωρισμός και από αυτού του, του θέματος. Γι' αυτό λοιπόν νομίζω ότι όλοι μας γνωρίζουμε ότι εφέτος ε, πρέπει να υπάρχει μια ε, πολύ δυναμική προσέγγιση ε, για να οριστούν τα απαραίτητα βήματα, το τι μπορούμε να κάνουμε χωρίς αλλαγές στις συνθήκες και το τι χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να σταθεροποιήσουμε την κατάσταση και πού χρειαζόμαστε και αλλαγές στις συνθήκες. Πάντως πρέπει να υπάρχει ένα σαφής ε, χάρτης πορείας, γιατί αλλιώς δεν θα μπορέσουμε να εκπληρώσουμε το καθήκον μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Συνσηγητά για την ομάδα S&D. Πολ Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Μου αρέσει δε αυτό το δικό χάρτη. Γιατί δεν ξέρουμε τι προβλήματα θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε στο μέλλον. Και καλό είναι να έχουμε μέσα για να προστατεύσουμε και να εξασφαλίσουμε το ευρώ. Και δεν είμαστε ακόμα εκεί. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι αυτό που μου αρέσει στην έκθεση είναι η ιδέα να δώσουμε κίνητρα για διαφορετικές μεταρρυθμίσεις. Είναι μια καλή ιδέα αυτή. Και εμείς πρέπει να την προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο. Δηλαδή να δούμε τον ενωσιακό προπολογισμό σε έναν τρόπο να δώσουμε κίνητρα για τα ευρωπαϊκά δημοσιογραφά θα μπορούσε να πει κανεί. Πώ συνεισφέρει μια χώρα σε ευρωπαϊκέ λύσει. Τέλο πάντων, θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε τι χώρε να υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν συγκεκριμένε πολιτικέ. Και βέβαια, αυτό δεν θα πρέπει να περιοριστεί ε, στο ESM ή στο μετασχηματισμό αυτού του μηχανισμού, αλλά να εφαρμόζεται στον προπολογισμό εν γέννη και να μην είναι απλά ένα μέσο ευρωπαϊκών πολιτικών, αλλά και για την αλληλεγγύη είναι κάτι πολύ σημαντικό. Γιατί είναι αμφίδρομη η αλληλεγγύη. Η Ευρώπη πρέπει να βοηθήσει τις χώρες να προβούν στις αλλαγές αυτές, αν θέλει βέβαια η Ένωση να γίνουν αυτές οι αλλαγές. Επίσης, για τη δημοσιονομική ικανότητα υπάρχουν τρεις πυλώνες, αυτά είναι σαφές. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσον θα πρέπει να αναλάβει όλες αυτές οι λειτουργίες, θα μπορούσε να περιοριστεί στα σύμμετρα ή συμμετρικά σοκ ή στη σύγκληση, αλλά αυτοί οι τρεις πυλώνες είναι απαραίτητοι για την προστασία του ευρώ. Βέβαια, εξακολουθούν να παραμένουν πολλά ερωτήματα. Δεν έχει ολοκληρωθεί ο δικός χάρτης, αν δεν τον συμβουλευτούμε μπορεί και να χαθούμε στο δρόμο. Πώς οι δημοσιονομικοί κανόνε μπορούν να συμβιβαστούν με τη δημοσιονομική ικανότητα. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Δεν μπορούμε να το αγνοούμε. Μπορούμε να κάνουμε περικοπές με βάση ε, του δημοσιονομικού κανόνε ε, και από την άλλη να μιλάμε για δημοσιονομική ικανότητα. Μου φαίνεται λίγο μπερδεμένο όλο αυτό. Και κάτι άλλο που προκαλεί σύγχυση είναι τι είναι εθνικέ αρμοδιότητε και ευθύνε και τι είναι ευρωπαϊκέ. Θα ήθελα λοιπόν οι δύο συνεισηγητέ να τα ξεκαθαρίσουν όλα αυτά. Σε ό,τι δεν αφορά τη σύγκληση, το να δώσουμε κίνητρα για τις διορτικές μεταρρυθμίσεις αρκεί ή και πού φτάνουμε, τι θέλουμε. Να πει, παραδείγματο χάρη, ξέρει στο Παρίσι τι εργασιακές μεταρρυθμίσει θα πρέπει να κάνει. Επίσης, η ευθύνη για τη δημοσιονομική πολιτική είναι στο εθνικό επίπεδο ή στο ευρωπαϊκό. Και αν είναι στο εθνικό είναι αποκεντρωμένη. Και αυτή η ρήτρα για τη μη διάσωση, το non-bailout. Περί πρόκειται. Δεν είναι σαφής η διάκριση εθνικού και ευρωπαϊκού επίπεδου. Άρα η γενική μου παρατήρηση είναι ότι δυσκολεύομαι να δω τι είναι εθνικό και τι είναι ευρωπαϊκό ως ευθύνη, ω καθήκον και αυτό όμως πρέπει να διευκρινίσετε, είναι σημαντικό. Υπάρχουν και κάποια άλλα σημεία που δεν είναι σαφή. Το πρώτο είναι πώς ένα εργαλείο της Ευρωζώνης ε, εντάσσεται στον ενωσιακό, στην ενωσιακή κοινοτική, όπως λέγαμε, μέθοδο. Δεν ξέρω, μήπω χρειάζεται μια διαδικασία λήψης αποφάσεων ένα κοινοβούλιο τη Ευρωζώνη. Αυτό δεν αναφέρεται στην έκθεση. Τέλο, η δημοσιονομική ικανότητα. πώ λαμβάνει υπόψη ή πώ εντάσσεται και πώ προσαρμόζεται με τον ευρωπαϊκό προπολογισμό και αντιμετωπίζει τα προβλήματα του ευρωπαϊκού προπολογισμού. Δηλαδή, για παράδειγμα, ότι τα κράτη-μέλη λένε ναι και δεν κάνουν τίποτα στην πράξη και άρα έχουμε καθυστέρηση πληρωμών πώς η δημοσιονομική ικανότητα θα μπορούσε τελικά να βοηθήσει για να εφαρμόζονται οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνω στο πλαίσιο του νησιακού προπολογισμού. Πάντως, ο δικός χάρτης χρειάζεται και πρέπει να τον επεξεργαστούμε. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Για την ομάδα ECR, κύριος Κόλμελ. Δεν είναι εδώ. Λένερ. Kiitos puheenjohtaja. Aluksi voin todeta, että... Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν ε, να πω ότι ε, σε μεγάλο βαθμό συμφωνούμε με τον κύριο Μιούρζαν και με τον ε, κύριο Μπάλτσε. Εδώ η βάση είναι το να έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία ε, χρησιμοποιεί τον προεπλογισμό της ε, για να ρυθμίσει θέματα που αφορούν ε, στα κράτη-μέλη. Κάτι τέτοιο βέβαια σημαίνει σύγκρουση ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτη-μέλη. Αυτό που επιθυμούμε είναι να υπάρχει ένας προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, που θα μπορεί να οδηγήσει σε μεταφορές ε, Αυτές οι μεταφορές ε, είναι δικαιολογημένες. Η δυνατότητα μεταφορών θα μπορούσε να οδηγήσει σε moral hazard ε, και όχι σε μεταρρυθμίσεις. Δεν νομίζω ότι κάτι τέτοιο μπορούμε να το εμποδίσουμε, παρότι αυτό αναφέρεται στην έκθεση. Οι διαφορές στην ανταγωνιστικότητα και στην παραγωγικότητα απλά είναι πολύ μεγάλες ε, ε, στην Ευρωζώνη. Και αυτός είναι ένας πολύ μεγάλος κίνδυνος. Επίσης, ε, στην έκθεση δεν γίνεται λόγος για πειθαρχία που πρέπει να υπάρχει στην αγορά. Δηλαδή, γίνεται λόγος ε, για την ε, ρεσιμότητα για προϋποθέσεις που θα συνδέονται με την αλληλεγγύη, αλλά αυτό είναι πάρα πολύ επιφανειακό. Οι διαθροτικές μεταρρυθμίσεις είναι πολύ δύσκολες και στη Φινλανδία. Η κυβέρνηση στη Φινλανδία αυτή τη στιγμή προγραμματίζει εκτεταμένες ε, μεταρρυθμίσεις ε, και περικοπές δημοσίων δαπανών. Ε, οι μεταρρυθμίσεις όμως παρότι βραχυπρόθεσμα πρόθεσμα μπορεί να μοιάζουν δύσκολες, μακροπρόθεσμα είναι απαραίτητες ένας μηχανισμός που ε, οδηγεί σε μεταφορές δεν είναι ευκταίος. θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας ε, για τη χρηματοδότηση, αλλά αυτό δημιουργεί πρόβλημα, γιατί ο ε, Μηχανισμός Σταθερότητας είναι ένα ταμείο για περίοδο, περίπτωση Κρήτης, οι διοκτήτες είναι τα κράτη-μέλη. Ως εκ τούτου το Κοινοβούλιο ε, δεν μπορεί να λάβει αποφάσεις για τα κονδύλια του ταμείου αυτού. Η πολιτική ομάδα των, ε, του ECR, τουλάχιστον για αυτά τα θέματα, θα καταθέσει τροπολογία. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς... Και τώρα θα θέλω να δώσω το λόγο ε, και την προεδρία στον Ζαν Ακτουή. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ τους δύο εισηγητές μας για αυτό το σχέδιο έκθεσης που συζητούμε σήμερα και είναι κρίσιμη η χρονική στιγμή. Όπως όλοι, έτσι και εγώ, σέβομαι το νομικό πλαίσιο. Αλλά, λαμβανομένης υπόψη της κατάστασης, θεωρώ ότι είναι άκρος απαραίτητο να έχουμε και ένα μια σαφή πολιτική εικόνα και ένα όραμα. Πού θέλουμε να πάμε δηλαδή. Όταν δημιουργήσαμε το νέο νόμισμα, είχαμε μια κοινή κυριαρχία αν θέλετε, την νομισματική κυριαρχία. Οι εθνικές κεντρικές τράπεζες ε, έγιναν μέτοχοι της ΕΚΤ και κατά κάποιο τρόπο ε, δημιουργήθηκε μια ομοσπονδιακή δομή, ένας ομοσπονδιακός θεσμός, αλλά δεν συναγάγαμε συμπεράσματα σε επίπεδο διακυβερνητικό, κυβέρνηση. Δηλαδή τότε η συζήτηση ήταν αν θα έπρεπε να δώσουμε βάρος σε έναν κανόνα, συνειδεκτίας αν θέλετε, να ορίζουμε κάποια όρια, ε, απαράβατα και όταν ε, τα υπερεύαιναν ε, αυτά τα όρια θα έπρεπε να επιβάλλονταν κυρώσεις στις χώρες που τα έπραταν ή αν θα έπρεπε να έχουμε μια οικονομική, δημοσιονομική κυβέρνηση. Στη συνθήκη του Άμστερνταμ καταγράφηκε η επιλογή μας για έναν κανόνα και ζητήσαμε από το Eurogroup που αποπαρτίζεται από τις υπουργούς οικονομικών των κρατών μελών της Ευρωζώνης να ασκούν τον έλεγχο και να αποφαίνονται για κυρώσεις. Από την αρχή μπορούμε να πούμε δηλαδή ότι δεν έγινε σεβαστός ο κανόνας, οι κυρώσεις δεν επιβλήθηκαν ποτέ δεν αναγγέλθηκαν καν και μετά από πάνω από 15 χρόνια Ευρωζώνης δεν επιβλήθηκε ποτέ καμία κύρωση, άρα ο κανόνα ή δεν υπάρχει, δεν εφαρμόζεται τέλο πάντων. Και η κυβέρνηση εξακολουθεί να μην υπάρχει. Άρα δεν υπάρχει χειρότερη κατάσταση, δεν υπήρξε σύγκληση και δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι και μια βέλτιστη οικονομική ζώνη, ευρωζώνη. Τώρα, αυτή η αρχή περί δημοσιονομικής ικανότητας Ευρωζώνης είναι κάτι επίκαιρο. Όπως λειτουργεί σήμερα η Ευρωζώνη, η πολιτική οικονομική δεν υπάρχει. Είναι η Ευρωζώνη μια προσθήκη εθνικών πολιτικών. Και η προσπάθεια που γίνεται είναι λίγο πολύ να συντονιστούν μεταξύ τους αυτές τις πολιτικές και ο δικητής της ΕΚΤΑ αναζητεί επιματέω έναν ε, κυβερνητικό διαμεσολαβητή και συνομιλητή για να προχωρήσει ένα πώληση μίξ. Δεν λειτουργεί λοιπόν σωστά η Ευρωζώνη. Εγώ αποδίδω μεγάλη σημασία στις προτάσεις των δύο εισηγητών, τους οποίους και συγχαίρω για τη φιλοδοξία, φιλόδοξη προσέγγιση. Δεν μπορούμε να μείνουμε ε, στην κατάσταση αυτή, γιατί η κατάληξη θα είναι πολύ άσχημη. Τώρα θα πρέπει να δούμε αν θα δημιουργήσουμε έναν ξεχωριστό προπολογισμό της Ευρωζώνης, διαφορετικό από τον ενωσιακό προπολογισμό, τον 28. Γιατί θα είναι πολύ δύσκολο να καταλάβουμε τι γίνεται. Ήδη ο προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και τόσο εύληπτος, σαφής, ιδίω μετά τα trust fund και τους ειδικού ε, οργανισμούς, τους δορυφωτικούς εκτελεστικούς οργανισμούς. Εμείς λοιπόν είμαστε υπέρ της διάκρισης των δύο προπολογισμών. Ένας ο ενωσιακός, άλλος ο προπολογισμό της Ευρωζώνης. Τώρα, πώς θα εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσαμε να φανταστούμε ε, περαιτέρω εισφορές ε, γιατί αυτό θα επιβάρει πολύ τους κατούς φορολογούμενους, αλλά θα μπορούσε να υπάρξει μια μεταβίβαση αρμοδιοτήτων. Παραδείγματο χάρη για την ε, ανεργία, το επίδομα ανεργία. Είναι κάποια παραδείγματα αυτά. Δείτε τι γίνεται με τον αμερικανικό προπολογισμό. Που είναι το 17-18% του ΑΕΠ πρώτα απ' όλα, τον είπα. Και το μισό είναι αφαιρωμένο σε κοινωνικές δράσεις, δράσεις αλληλεγγύης. Θα μπορούσαμε ίσως να φανταστούμε σε ό,τι αφορά την Ευρωζώνη μία μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους τομείς αυτούς. Δηλαδή η χρηματοδότηση να γίνεται από μία μεταφορά πιστώσεων, πόρων, τα κράτη-μέλη δηλαδή δεν θα έφερναν, δεν θα επομίζουν πλέον αυτό το βάρος και αυτά τα χρήματα θα πήγαιναν στον ε, προπολογισμό της Ευρωζώνης. Βέβαια αυτός ο προπολογισμό σίγουρα θα πρέπει να βοηθήσει στην ενεργοποίηση διαφορετικών μεταρρυθμίσεων και στη σύγκληση των νομοθεσιών για να μπορέσει η Ευρωζώνη να γίνει βέλτιστη και ίσως και με έναν Υπουργό Οικονομικών ε, που δεν θα τον κατηγορεί κανείς για σύγκρουση συμφερόντων, δεν θα είναι δηλαδή Υπουργός Οικονομικών σε μια χώρα της Ευρωζώνης και ένα ε, ταμείο αν θέλετε, δημόσια ταμείο της Ευρωζώνης. Και εδώ θα σταματήσω. Ε, Ρομπέρτο νομίζω μου έδωσες και την Προεδρία. Ωραία. Άρα να δώσω τον λόγο τώρα στον Νίλς Τόρβαλς και μετά στην Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχά, θα ήθελα να ευχαριστήσω <clears throat> τους εισηγητέ, συνεισηγητέ για την εργασία τους. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι περισσότερα ερωτήματα κατέγραψαν από ότι θα μπορέσουμε να απαντήσουμε στη διάρκεια αυτής της συζήτησης και κατά κάποιο τρόπο αυτό είναι καλό διότι όντως έχουμε πολλά προβλήματα μπροστά μας και πρέπει να βρούμε τον τρόπο να το διορθώσουμε. Ακόμα και αν για να φτιάξει κανείς ένα οδικό χάρτη από αυτό, ε, εξόδου από αυτό το μπέρδεμα θα είναι πολύ δύσκολο. Είναι ευκολότερο να κάνει κανείς τα πράγματα εκ των προτέρων παρά εκ των υστέρων. Όλα τα προβλήματα αυτά είχαν ληφθεί υπόψη πριν να φτιαχτεί η Ευρωζώνη τότε μάλλον θα ήταν τώρα ευκολότερο να ήμασταν σήμερα εδώ. Το να διορθώσουμε τα πράγματα όπως πρέπει σήμερα να κάνουμε είναι πολύ δυσκολότερο. Να σας δώσω κάποια παραδείγματα για τις αμφισημίες τις οποίες έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Μιλάμε πολύ σε αυτό το έγγραφο για συμμετρικά σοκ. Αν επανέλθουμε στη θεωρία του Μαντέλ, ε, να είστε βέβαιοι ότι Όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα συμμετρικό σοκ, στη συνέχεια όλα ομαλοποιούνται. Αλλά βέβαια αυτός ήταν ένας αισιόδοξο ε, της δεκαετίας του 80. η σημερινή πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική. Ορισμένε χώρε έχουν να αντιμετωπίσουν πολύ έντονα ασυμμετρικά σοκ λόγω του ότι τι χτύπησαν οι καινοτομίε με διαφορετικού τρόπου και η πραγματικότητα του οικονομικού κόσμου τους χτύπησε με διαφορετικού ε, τρόπου. Γι' αυτό και φαντάζομαι ότι θα έχουμε να ζούμε με τα ασυμμετρικά κύματα σοκ καθ' όλη τη διάρκεια του αιώνα. Και θα πρέπει να προσαρμοστούμε σε αυτό. Αλλά ταυτόχρονα αυτό προκαλεί πολλά ερωτήματα. Πώς θα φτιάξουμε ένα σύστημα το οποίο να είναι ανθεκτικό απέναντι σε αυτά τα συμμετρικά σοκ. Ένα άλλο πρόβλημα που έχουμε, μάλλον αφησιμένο, είναι ο τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται η συνοχή σε, αυτό, αυτή την έκθεση. Να σα δώσω ένα παράδειγμα. Εάν πούμε ότι η πολιτική συνοχή έχει αποτύχει, μάλλον ε, μιλάμε για δύο διαφορετικέ προσεγγίσει. Ε, το θέμα είναι ότι η συνοχή έχει αποτύχει. Αν δούμε τις στατιστικές, η συνοχή δεν έχει λειτουργήσει χονδρικός από το 1975 και έκτοτε. Ε, μάλλον δεν καταφέραμε να τηρήσουμε τη συνοχή. Μάλλον δεν καταφέραμε να διαπιστώσουμε την αποτυχία τα τελευταία 40 ε, χρόνια. Όταν λέμε όμως ότι η πολιτική συνοχή έχει αποτύχει, τότε ε, προσκρούμε σε ένα πιο σοβαρό πρόβλημα, γιατί λέμε ταυτόχρονα ότι η πολιτική συνοχή θα έπρεπε να έχει πετύχει κάτι περισσότερο από αυτό που επέτυχε. Και άρα σημαίνει ότι υπάρχουν περισσότερες δυνατότητες από την πλευρά της πολιτικής. Δηλαδή οι πολιτικοί απέτυχαν. Και εδώ έρχομαι τώρα στο ζήτημα του ηθικού κινδύνου, moral hazard. Μάλλον θα είδατε στις εφημερίδες πριν από λίγες μέρες ότι οι Έλληνες πολίτες χρωστούν στο κράτος τους 8 δισεκατομμύρια μη καταβληθέντων φόρων. Και αυτό είναι ένα από τα κεντρικά προβλήματα ε, της ε, ελληνικής κρίσης χρέους. Δεν πληρώνουν τους φόρους τους. Άρα λοιπόν εδώ προκύπτει πρόβλημα ηθικού κινδύνου. Είναι καλό λοιπόν που έχουμε αυτή την έκθεση, διότι όντως ε, δακτυλοδείχνει διάφορα σημεία που έχουμε και προβλήματα που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι δεν υπάρχουν εύκολες απαντήσεις αν ε, λάβουμε υπόψη ότι έχουμε περίπου μια εβδομάδα για να βρούμε καλή λύση για όλα αυτά, τότε να πω συγχαρητήρια στους εισηγητές, συγχαρητήρια στους σκιώδεις, γιατί τις επόμενες μέρες θα περάσετε ε, από φωτιά και σίδερο και αξίζετε τα συγχαρητήρια εκ των προτέρων. Ευχαριστώ. Η κυρία Νεριέντα δεν είναι εδώ, ούτε ο κύριος Δεμάση από την ΚΟΕ, ο κύριος Μαραγάλ ούτε, αλλά ο κύριος Μπάς μας ο Μπάς μας ακούει, έχει και το λόγο. Κάνατε εξαιρετική δουλειά. Σας συγχαίρω. Ε, είναι πολύ καλό σημείο κίνηση για να συζητήσουμε τις ε, συνέπειες ή τα διάφορα μέρη όλου αυτού του μπερδέματος. Νομίζω πως είναι καλή βάση λοιπόν για να ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις και εδώ θέλω να ευχαριστήσω τους εισηγητές που το κατάφεραν αυτό ε, γνωρίζοντας ότι προέρχονται από διαφορετικές χώρες και διαφορετικές πολιτικές ε, συνιστώσεις το να μπορέσουν να συντάξουν μια τέτοια έκθεση ήδη ήταν ε, εξαιρετικό επίτευγμα και ελπίζω ότι και στις ομάδες σας θα σας στηρίξουν σε αυτά που προσπαθείτε να πετύχετε. Εν τέλει, βασικά αυτό που θέλουμε να δούμε είναι πώς θα βρεθεί η ισορροπία ε, μοιρασιά του κινδύνου αλλά και της κυριαρχίας. Από τη στιγμή όμως που έχουμε κοινό νόμισμα χρειαζόμαστε να έχουμε και ε, ε, δημοσιονομικές δυνατότητες. Ίσως κάποιοι ακόμα να το αρνούνται, αλλά είναι γεγονός ότι δεν μπορούμε να μην έχουμε δημοσιονομικές δυνατότητες από τη στιγμή που έχουμε κοινό νόμισμα. Αν δω τους τρεις πυλώνες τώρα, να πω καταρχάς ότι η έκθεση φαίνεται να βασίζει τις υποθέσεις στο ότι ο μηχανισμός σταθερότητας είναι ο μοναδικός μηχανισμός που υπάρχει. Και αν δούμε ποιες είναι οι προσδοκίες από αυτόν τον μηχανισμό, πιστεύω πως περιμένουμε υπερβολικά πολλά από αυτό. Και αυτό θα πρέπει να το προσέξουμε και θα πρέπει να δούμε και άλλες δυνατότητες χρηματοδότηση από αυτόν και μόνο το μηχανισμό γιατί αυτή η έκθεση τουλάχιστον για το σημερινό πλαίσιο βασίζει πολλές ελπίδες αποκλειστικά στον ESM. Ε θα ήταν καλό επίση να ρωτήσουμε από τι νομικέ υπηρεσίε να μα δώσουν πληροφορίε για το σε ποιο βαθμό είναι δυνατόν να έχουμε και κάποιον άλλο, κάποιο άλλο μέσο εκτό από το ESM με βάση τις ισχύουσες συνθήκε. Γιατί πιστεύω ότι αν όλα τα βασίσουμε σε αυτόν τον μηχανισμό θα έχουμε προβλήματα ασυμμετρικά σοκ για αντιμετώπιση του, Ενώ από τα πιο σημαντικά ζητήματα για τη δική μα ομάδα θα είναι ότι εδώ πρέπει να είναι αυτόματη αυτόματος σταθεροποιητής και δεν θα χρειάζεται να σωρό πολιτικά κριτήρια να ισχύσουν πριν ε, να, ε, να, να μπει σε εφαρμογή αυτό, αυτή η αντιμετώπιση των ασυμμετρικών σοκ. Γιατί ε, αν χρειαστεί να περάσει πολιτική διαδικασία, θα καθυστερήσει. Θα πρέπει αντίθετα να γίνεται αυτόματα και οι δείκτες, οι όροι να έχουν προκαθοριστεί να μην περιμένουμε να τους καθορίζουμε στη διάρκεια μιας κρίσης. Γιατί ο κενό χρηματοδότησης, ή πάση περιπτώσει το μέσο το επενδυτικό, για μας είναι σημαντικό κατά κάποιο τρόπο η Ευρώπη να έχει ένα, έχει μάλλον ένα ευρύτερο επενδυτικό κενό και δεν θα λυθεί το πρόβλημα μόνο με αυτή την προσπάθεια. Πρέπει να δούμε την δυνατότητα να ανανεώσουμε το εύση που υπάρχει αλλά που δεν λειτουργεί φούλα αν δούμε τις επενδύσεις. Επίσης, ε, κατά ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να δώσουν ε, input, χρήματα σε αυτή τη, το πυλώνα της σύγκλησης. Αλλά σε ποιο βαθμό, αν τα κράτη-μέλη αυτό δεν το καταφέρουν, θα μένει εν λειτουργία αυτός ο πυλώνας της σύγκλησης. Και εδώ λοιπόν πρέπει να σκεφτούμε άλλους μηχανισμούς απόδοσης, ε, ανταμοιβή, ώστε να εξασφαλίσουμε ότι τα, μέλη, τα μελη θα συμμετέχουν. Αυτές είναι οι δικές μας ιδέες, τις προτείναμε στη διαπραγμάτευση ε, Νίλς, ε, περιμένω. Δεν ξέρω εσύ αν το περιμένεις με τόση ανυπομονησία. Δεν το κατάλαβα ακριβώ από αυτά που είπες. Και πιστεύω ότι από αυτές τις βάσεις θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα θέση τελικά ως Κοινοβούλιο, ώστε να εξασφαλίσουμε ότι η συζήτηση θα διευρυνθεί. Γιατί το να έχουμε εδώ μια θέση, εντάξει, αλλά η πιο σημαντική συζήτηση θα πρέπει να γίνει με τα κρατημέλη. Και αυτή είναι η μεγαλύτερη πρόκληση ως Κοινοβούλιο, αν θα μπορέσουμε σε αυτό να παίξουμε ρόλο. Και πάλι ευχαριστώ λοιπόν τους συνεισηγητές για την ε, θέση τους. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μαραγκάλ κατέφτασε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Με κίνδυνο ε, να πω πράγματα που, δεν, που έχουν ήδη υποθεί, γιατί έλειπα ε, και θα μιλήσω στα ισπανικά όπως πάντα. Πρώτον, δεν άκουσα όλες τις παρεμβάσεις. Βέβαια, όπως είναι προφανές. Οπότε, ίσως να επαναλάβω κάποια πράγματα. Πάντως ε, συμφωνώ με τα όσα είπε ο συνάδελφος μόλις. Ε, δεύτερον, πιστεύω όχι μόνο την καλή ευκαιρία, αλλά πρόκειται για ένα καλό έγγραφο επί το οποίο να εργαστούμε για να αποτελέσει δηλαδή τη βάση για τη θέση του Κοινοβουλίου. Πρόκειται για προβληματισμό που ταιριάζει με το ρόλο που μπορεί να παίξει το Ευρωκοινοβούλιο σε αυτό το θέμα που είναι τόσο περίπλοκο και ε, είμαστε στη μέση ε, συμπίπτη με τη συζήτηση του PDP ε, αλλά ταυτόχρονα αναλαμβάνουμε και ευθύνη για να δώσουμε ορισμό και περιεχόμενο στο τι πρέπει να είναι η Ευρωζώνη, η διακυβέρνησή της, οι μηχανισμοί της και οι δυνατότητες ε, ε, εφαρμογή όλων αυτών. Έχω τέσσερα ζητήματα να θίξω. Το ένα είναι θετικό. Θα πρέπει ως ομάδα αλλά και ως κοινοβούλιο να βασιστούμε σε αυτό το κείμενο. Υπάρχει όμως ένα θέμα πιο, πιο συγκεκριμένο, μια πιο προσωπική μου άποψη είναι ότι υπάρχει μια αμφισημία ε, όσον αφορά τα συμμετρικά και τα συμμετρικά σοκ. Ε, γιατί τα συμμετρικό σοκ είναι μια συμμετρία αντιθέτων ε, συστημάτων που δεν μπορούμε να αντιδράσουμε καλά. Έχουμε ελληματικούς χρεώστες από τη μια πλευρά, και δεν μπορούν να ξεπεράσουν μια συγκεκριμένη κατάσταση και έχουμε την κατάσταση των πιστωτών από την άλλη πλευρά. Είναι το αντίθετο από αυτό που συνήθως αντιμετωπίζουμε δηλαδή. Θα πρέπει αυτό να το έχουμε υπόψη μας για να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα μέσα στο πλαίσιο αυτής της ασυμμετρικής σημειολογίας που περιλαμβάνεται σε αυτή την έκθεση. Και αυτό για να μπορέσουμε να το συνδέσουμε με τα υπόλοιπα, γιατί σε ολόκληρη την έκθεση θα πρέπει κάτι να συμπληρώσουμε, ότι δηλαδή οι τρεις πυλώνες που μπορούμε να θεωρήσουμε, να τους εξετάσουμε μόλις, μάλιστα χωριστά και να συμφωνήσουμε για τον προορισμό, για το περιεχόμενο γενικά, όμως επιπλέον θα πρέπει να ε, συνδέονται μεταξύ τους καταλήλως, γιατί διαφορετικά, όπως συχνά συμβαίνει σε αυτούς τους θεσμούς, υπάρχει ο κίνδυνος να προχωρήσουμε, αλλά χωριστά. Το καθένας, ο καθένας στο δρόμο του, ο καθένας να έχει τη λογική του, το μέσο του, τους στόχους του, αλλά που τελικά να μην συναντώνται. Πρέπει δηλαδή να ε, υπάρχει εκ των προτέρων ορισμός ε, διασύνδεσης των τριών πυλώνων. Επίσης, ε, από το building mechanism να περάσουμε σε έναν Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο είναι μια καλή ιδέα. Το θέμα είναι πόσο αυτό θα συνδεθεί με τους υπόλοιπους στόχους και τις υπόλοιπες πολιτικές συμπεριλαμβανομένες της διαχείρισης των ε, ανισορροπιών. Τώρα, το Ταμείο Χαλιπών Καιρών και η ε, ασφάλεια ανεργίας επίσης είναι πολύ θετικά μέσα. Αλλά θα πρέπει να τους προσθέσουμε και κάποιο αιρεσιμότητα, κάποιους όρους, κάποιες ευθύνες, γιατί διαφορετικά θα μπορεί εδώ να καλύπτεται η μόνιμη διαφάνεια και το moral hazard. Θα πρέπει να είμαστε πιο φιλόδοξοι και πιο συγκεκριμένοι σε αυτή την κατεύθυνση. Λοιπόν, αιρεσιμότητα για το Ταμείο Χαλεπών Καιρών και την ασφάλεια ανεργίας. Στην έκθεση, και εδώ μπορούμε να συζητήσουμε και να συμφωνήσουμε νομίζω, λείπει αυτό που μόλις ακούσαμε, ότι έχουμε δηλαδή ένα τραπέζι με, με δυο πόδια, αλλά λείπει και το πόδι των επενδύσεων. Άμα δεν έχει και ένα τρίτο πόδι επενδύσεις, το τραπέζι δεν θα σταθεί. Δεν θα έχουμε ένα πλήρες πακέτο και τη σχέση ανάμεσα σε όλα αυτά που θα επιτρέψει να ορίσουμε ευρωπαϊκές πολιτικές στην κατεύθυνση της απασχόλησης, της ισορροπίας ε, και της ε, σύγκλησης ανάμεσα σε όλα τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό λοιπόν το τρίτο πόδι, δηλαδή επενδύσεις, επενδύσεις δημόσιες, ευρωπαϊκές επενδύσεις με ευρωπαϊκούς μηχανισμούς διαχείρισης τους αλλά και ανάθεση των κονδυλίων και έλεγχος από πλευράς των κρατών μελών. Και το τέταρτο θέμα, το τέταρτο σχόλιο που έχω, που είναι στην έκθεση και τελειώνω, Πρόεδρε, είναι το θέμα της διακυβέρνησης, όπου υπάρχει λεπτή ισορροπία ανάμεσα στην Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, δημοσιονομικές δυνατότητες για την Ευρωζώνη και ευρωπαϊκός προϋπολογισμός. Και αυτό θα πρέπει να το λύσουμε. Και η έκθεση αυτή μας λέει ότι ναι, πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε ε, για να βρούμε την κατάλληλη διατύπωση και για αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε, και εγώ σας ευχαριστώ. Και τώρα το λόγο έχει ο Μάρκο Βάλλη. Πρόεδρε, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ζητήσω ε, συγγνώμη από το συνάδελφό μου γιατί είχε ένα μικρό πρόβλημα υγείας και δεν μπορούσε να έρθει και θα παρέμβω εγώ. Λοιπόν, κοιτάξτε, η έκθεση τη διάβασα και κυρίως σε αυτά που έχουμε ορίσει. Ε, εγώ πρέπει να σας πω ότι δεν έχω πιστεί καθόλου. Ούτε η ομάδα μου έχει πιστεί. Ε, και διότι ε, από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει κανενός ε, είδους δημοκρατική επιλογή, τουλάχιστον από τις επιλογές που προτείνονται. Είναι επιλογές ε, οι οποίες έχουν γίνει από γραφειοκράτες, από εκπροσώπους συμφερόντων. Άρα δηλαδή οι άνθρωποι, οι απλοί άνθρωποι, όπως και εγώ, είμαστε αντικείμενο όλων αυτών των αποφάσεων και γι' αυτό θέλουμε να αντιδράσουμε. Το επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά. Βλέπω ότι Μιλάμε και πάλι για, με τις Νάλφο Μπέρες ε, για την έκθεσή της, για την έκθεση την οποία είχαμε ήδη ψηφίσει πέρσι. Έχουμε λοιπόν ένα νόμισμα το οποίο συνδέει 19 κράτη, το οποίο όμως είναι βαθιά ε, διαφορετικά μεταξύ τους ε, και γι' αυτόν τον δρόμο λόγο δημιουργούνται ανισορροπίες προσπαθούμε να λύσουμε το θέμα να υπάρχει ένας προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου τα κράτη-μέλη δίνουν τη συνεισφορά τους και θέλουμε να έχουμε έναν υπερυπουργό οικονομικών αλλά αυτό δεν είναι δημοκρατικό, θα επιβάλλει τα μεταρρυθμίσεις όπως στη Γαλλία βλέπουμε τι γίνεται, βλέπουμε τι έγινε στην Ιταλία και στην Ελλάδα καμία δημοκρατία, όλα θα επιβάλλονται ε, θα ξεπουληθούν τα κράτη, θα υπάρχουν ταμεία για να δανείζουν χρήματα και να πληρώνει κανεί ή να πληρώνουν τα κράτη ε, τα, τους τόκους. Αυτά λοιπόν επιβάλλονται με αυτό το πλαίσιο και δεν είναι κάτι το εφιές ε, που θα μπορούσε να χρησιμεύσει ε, τουλάχιστον για τη Γερμανία και την ε, Ολλανδία για να λειτουργήσει το ευρώ. Γιατί για να λειτουργήσει το ευρώ πρέπει οι χώρες που πλουτίζουν λόγω του ευρώ, οι χώρες αυτές να κάνουν επενδύσεις, να μεταφέρουν κονδύλια σε καθυστερημένες περιοχές και σε εξόχως απόμακρες περιοχές. Βλέπουμε όμως ότι δεν συμβαίνουν όλα αυτά, άρα δηλαδή το να προχωρήσει αυτό το σχέδιο σχέδιο, τουλάχιστον κατά τη δική μας την άποψη, δεν έχει νόημα. Γιατί δεν είναι δημοκρατικό, δεν είναι σωστό, γιατί δεν ε, έχει καμία καλή βάση. Αυτά πρέπει να τα πούμε ξεκάθαρα. Ε, κατόπιν τούτου, όσον αφορά το θέμα της μεταρρύθμισης των συνθήκων, για να γίνεται σεβαστή η δημοκρατία και για να μπορούν να εφαρμοστούν διαφορετικές πολιτικές από αυτέ που επιθυμούν οι κερδοσκόποι ή τα μεγάλα συμφέροντα, για να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει στις συνθήκες να υπάρχει δυνατότητα opting out ε, για το ενιαίο νόμισμα. Δηλαδή να μπορεί κανείς να αποφύγει πολιτικές ε, προεκτάσεις λόγω του ενιαίου νομίσματος. Αυτό είναι δημοκρατικό. Άρα δηλαδή ένα δημοκρατικό μέτρο στις συνθήκες που θα επιτρέπει σε ένα κράτος και στους πολίτες να βγουν από μια παγίδα η οποία θα επιτρέπει ε, να εφαρμόζονται άλλες πολιτικές από αυτές των μεγάλων συμφερόντων. Αυτό θα ήταν ε, ιδιαίτερα ευτυχές. Είμαι, λυπάμαι που μόνος ε, που δεν μιλάω όπως όλοι οι άλλοι αλλά πρέπει να σας πω ότι είμαστε αρκετοί και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι το δικό μας το μέτωπο ε, στηρίζεται και τρέφεται από αυτή την αντίδραση. Να γίνεται σεβαστή η δημοκρατία, να λαμβάνονται δημοκρατικές αποφάσεις. Και αυτό το πλαίσιο που θέλετε να μας επιβάλλετε δεν είναι δημοκρατικό. Ε, θα αποφασίζονται όλα από γραφειοκράτες ε, και από ευρωβουλευτές όμως οι οποίοι δεν θα εξυπηρετούν τα συμφέροντα των απλών πολιτών. Σα ευχαριστώ. Εδώ είμαστε για να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Αυτό σίγουρα είναι δημοκρατικό. Έχουμε ακούσει τώρα όλους τους κοιόδες που είναι παρόντες και τώρα περνάμε στο Κατσεδιάι. Δεδομένου ότι πρέπει να επιστρέψουμε αυτή την, την αίθουσα οπωσδήποτε στις 16.30 στην Επιτροπή ΕΚΟΝ. Ναι, θα πολύ, να, να, είσαι πολύ αυστηρός. Το λόγο έχει ο Ροπέρτο Γουαλτιέρη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ δεν θα επεκταθώ όσον αφορά την αναγκαιότητα της, ε, των δημοσιονομικών δυνατοτήτων, γιατί είπαμε ότι πρέπει να υπάρχει ένας ε, προϋπολογισμός για την ενιαία αγορά και για τις τρεις, ούτε και τους τρεις πυλώνες, γιατί η γνώμη μου έχει οριστεί έχει, είναι ήδη γνωστή όσον αφορά την αντιμετώπιση και απορρόφηση συμμετρικών και συμμετρικών σοκ. Θέλω να κάνω μόνο κάποιε παρατηρήσει για τον κύριο Μούρασεν και για τι παραγράφου 9 και 19 τη έκθεση, γιατί πρέπει να αποφύγουμε τι παρεξηγήσει. Έχουμε εδώ δύο διαφορετικά πράγματα. Έχουμε το ρόλο του μηχανισμού σταθερότητα και την πιθανή του ένταξη στη συνθήκη και την πιθανή εξέλιξή του προ έναν Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο. Πολύ ωραία φιλοδοξία αυτή Άλλο ένα είναι η δημιουργία των δημοσιονομικών δυνατοτήτων και το, η ένταξη αυτών στο ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο. Για, αυτά είναι, ε, συνδέονται, αλλά, γιατί το ESM είναι ένα εργαλείο, είναι ένα μέσο, αλλά εδώ εγώ διαφωνώ με τον κύριο ότι η αλλαγή συνθήκη είναι η, η μόνη προϋπόθεση. Ναι, βεβαίως μια αλλαγή της συνθήκης θα σήμαινε πιο ρεαλιστική τη λύση, αλλά δεν είναι η μοναδική δυνατότητα που έχουμε. Γι' αυτό θέλω να τονίσω ε, ότι το άρθρο 175.3 ε, της συνθήκης είναι εξαιρετική νομική βάση και το 116.7 που ορίζουν ότι η συγκεκριμένη λειτουργία δεν είναι ε, προκαθορισμένη. Χρησιμοποιήθηκε, ας πούμε, για το σχέδιο Juncker. Είναι εξαιρετική νομική βάση και όσον αφορά την ένταξη στον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό έχουμε το άρθρο 21 του δημοσιονομικού κανονισμού που ορίζει σαφώς ότι μπορείς να εισάγεις ε, συγκεκριμένες γραμμές του προϋπολογισμού εντός του προπολογισμού και δεν απαιτείται ούτε καν η ομοφωνία για τους ίδιους πόρους ε, υπό το 3.11.3. Θα ήταν ακόμα μια δυνατότητα. Έχουμε λοιπόν διάφορες δυνατότητες σύμφωνα με τις ισχύουσες συνθήκες για συγκεκριμένο γραμμή του προπολογισμού. Υπήρχε νομική βάση και στο η πρόταση CCI της Κομισιόν, την αρχική πρόταση. Για το συντονισμό τώρα έχουμε το άρθρο που αφορά την διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών. Αυτά όλα θα μπορούσαν ήδη να χρησιμοποιηθούν. Θα είχαμε το 175 και το 136 και να έχουμε έναν ε, κώδικα σύγκλησης. Μετά έχουμε το θέμα του ESM και του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου που είναι πιο περίπλοκα. Εδώ υπάρχει συζήτηση αλλαγή για τις συνθήκων. Και αν θέλουμε να έχουμε έναν οδικό χάρτη θα πρέπει να ξεκινήσουμε βλέποντας τι μπορούμε να κάνουμε ήδη από τώρα εφόσον υπάρχει πολιτική βούληση. Γιατί όταν υπάρχει βούληση υπάρχει και ο τρόπος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο συνάδελφο Βεν Βάιζέκερ. Ναι, ευχαριστώ κύριε Αρτουή. Ήθελα να συγχαρώ τους δύο συνεισηγητές. Θεωρώ ότι είναι πολλά υποσχόμενο αυτό το σχέδιο έκτησης και το ζήτημα είναι πολύ δύσκολο. Και εντυπωσιάστηκα, γιατί ξέρω πόσο δύσκολο είναι να καταλήξει κανείς ένα τόσο καλά διαρθρωμένο έγγραφο. Βέβαια, για να καταλήξουμε σε ένα σημείο που και εδώ, στο Κοινοβούλιο, αλλά και πιο πέρα, θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε μια συζήτηση, θα πρέπει να ορίσουμε κάποια πράγματα. Κάποιες φορές γνωρίζω ότι χρειάζεται και η ασάφεια, αλλά δεν θα πρέπει πιο αναλυτικά και για τους τρεις πυλώνες να δούμε ποια είναι η ισορροπία μεταξύ ευθύνης και αλληλεγγύης. Δηλαδή να δούμε τι ακριβώς συνιστά εθνική ευθύνη στο δικό σας μοντέλο, τι είναι ευρωπαϊκή ευθύνη ή αρμοδιότητα γιατί πιστεύω ότι αυτό θα βοηθήσει πολύ και στο ίδιο πνεύμα. Καλό είναι να διευκρινίσουμε με αυτούς τους τρεις πυλώνες ποιοι είναι οι περιορισμοί στους εθνικούς για το μέλλον και πόσο ε, αξιόπιστοι θα είναι οι προπολογισμοί, ιδίως και με βάση τόσο είπε ο Επίσης θα μπορούσε να συζητηθεί περισσότερο το θέμα των επιλογών χρηματοδότησης για αυτή τη δημοσιονομική ικανότητα. Εσείς ε, μιλήσατε για τις δυνατότητε του ESM, αλλά νομίζω ότι θα μπορούσατε να αναφέρετε πιο αναλυτικά τις επιλογές. Είναι πολύ λεπτό το θέμα βέβαια Νομίζω ότι ίσω να ήταν ανεδαφικό να περιμένουμε κάτι περισσότερο, αλλά νομίζω ότι συστηματικά θα ήταν καλό να ε, εξηγείτε περισσότερο τι υπολογίε και για του διαφορετικού ε, πυλώνε, τι διαφορετικέ επιλογέ που μπορεί να είναι πλέον κατάλληλε σε κάθε περίπτωση. Τέλο, και επειδή έχουμε συζητήσει ω ένα βαθμό και το ζήτημα του τι μπορεί να γίνει χωρί αλλαγή συνθήκη και για το τι πρέπει να γίνει με αλλαγή συνθήκη, νομίζω ότι η αξιοπιστία του όλου αυτού οικοδομήματος έχει πολύ μεγάλη σημασία τόση, ώστε ίσως ορισμένα πράγματα δεν θα έπρεπε να τα κάνουν χωρίς αυτή τη συνθήκη. Και θα έπρεπε να πούμε ότι σε κάποια σημεία θέλουμε να είμαστε αξιόπιστοι, πρέπει να προβούμε σε αλλαγές της συνθήκης. Όχι αυτό το σύστημα της κοινής ευθύνης που έχουμε μέχρι τώρα, γιατί έχει λείψει προφανής αυτό το σύστημα. Δεν έχουμε πάρκει αξιοπιστία σε ορισμένου τομεί. Θα μπορούσαμε να έχουμε έδωση κοινή κυριαρχία για κάποια ε, σημεία, για κάποιου δημοσιονομικού περιορισμού. Αυτέ είναι οι παρατηρήσει μου. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Φερνάνδη το έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εισηγητές για τους ε, για τις προσπάθειές τους Μπέγκη και Περές είναι ένα καλό αρχικό έγγραφο ως βάση συζήτησης για να δούμε πώς θα οικοδομήσουμε αυτόν τον δημοσιονομικό πυλώνα ιδίως για την Ευρωζώνη. Ακούμε εθνικιστικές κορώνες ε, όμως ε, ότι δεν υπάρχει διαφάνεια, μιλάμε για τη δικτατορία των τεχνοκρατών των Βρυξελών, όμως αυτή η συζήτηση σαφώς δείχνει ότι υπάρχει διαφάνεια και λειτουργεί δημοκρατικά ε, η ευρωπαϊκή οικοδόμηση. Εγώ δύο σχόλια έχω να κάνω, διότι η έκθεση θεωρώ ότι είναι πολύ καλή και συνθέτει πολύ καλά τις προτάσεις για τους τρεις αυτούς πυλώνες. Σε αυτή την έκθεση πάντως καλό θα ήταν να συζητήσουμε τουλάχιστον το πώς θα εξασφαλίσουμε τη χρηματοδότηση. Είναι ένα ζήτημα που συζητείται Καλό είναι όμως να σκεφτούμε πώς θα χρηματοδοτηθούν αυτοί οι τρεις πυλώνες. Θα ήθελα να υπενθυμίσω, γίνεται και στην έκθεση το ίδιο, ότι υπάρχει αυτός ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας που δημιουργήθηκε το 2010. Αλλά νομίζω ότι κοιμάται τον ύπνο του δικαίου έκτοτε. Δηλαδή δεν του δίνεται ιδιαίτερη προσοχή. Πάνω όμως από 40 δις ευρώ είναι η δημοσιονομική του ε, ικανότητα και θα μπορούσε με το σχέδιο Juncker κατά κάποιο τρόπο να συνδυαστεί ή ίσως στο πλαίσιο αυτού του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ινστιτούτου προτείνει έκθεση αυτά τα 40 δις αποθεματικού που είναι στον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αυτό είναι η διαφορά με το τρέχον ε, σύστημα μπορούσε αυτά τα 40 δις ε, να χρησιμοποιηθούν Θέλουμε να βάλουμε τον ISM στο κοινοτικό και εκτιμενο στο κοινοτικό σύστημα. Αυτά τα 40 δις όμως θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση κεφαλαίου για αυτό τον μηχανισμό. Θα μπορούσαμε δηλαδή κατά κάποιο λόγο, de facto και de jure, να θεσμοθετήσουμε αυτόν τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητα που θέλουμε να χρησιμοποιηθεί ω βάση για αυτό το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο. Και έτσι αξιοποιήσουμε αυτά τα 40 δι, επαναλαμβάνω. Και σε άλλε συναντήσει έχουμε συζητήσει την έκτα. Μιλάμε για ίδιους πόρους μέσα στην Ευρωζώνη. Υπάρχει καλύτερος ίδιος πόρος μέσα στην Ευρωζώνη από αυτά τα κέρδη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Υπάρχει ένα άνθρωπο που θα μπορούσε με την, νομοθετική, την κανονική νομοθετική διαδικασία να τροποποιηθεί χωρίς να χρειάζεται μια επίσημη αλλαγή των συνθήκων για να δούμε ποια είναι η νομική βάση ώστε από το καταστατικό της έκτη να δούμε πώς μπορούμε το 20% των κερδών ε, να το διασώσουμε κατά κάποιο τρόπο για να μπορούμε να ε, δώσουμε ένα κομμάτι αυτών των κερδών ε, για τον προϋπολογισμό με την, τακτική, με την κανονική νομοθετική διαδικασία. Το λέει και το καταστατικό στο άρθρο 33.1α, το λέει και η συνθήκη της Λισαβόνας. Και έχουμε και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Οικονομικής Σταθερότητας που θα μπορούσε στο κεφάλαιο του ESM να δώσει κάποια χρήματα, κάποια κονδύλια για να μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε, όπως είπα, τους τρεις πυλώνες που είναι και το ζητούμενο. Ευχαριστώ, Σιλβί Κουλάρ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Να συγχαρώ και τους εισηγητές μας έχουν δώσει μια πολύ καλή βάση εργασία. Σε τρία σημεία θέλω να επιμείνω. Το πρώτο είναι ότι νομίζω ότι στόχος θα πρέπει να είναι αυτό που είπατε να γίνει βέλτιστη η λειτουργία της ε, Ευρωζώνης. Δεν το κάνουμε έτσι απλά και μόνο για να ευχαριστήσουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά για την καλύτερη χρήση των πόρων και του ευρώ ως ε, νομίσματος, που θα έπρεπε να φέρνει ευημερία. Και αυτή είναι η αρχή που θα πρέπει να μας διέπει. Δηλαδή, στόχος είναι να βελτιώσουμε τη λειτουργία της Ευρωζώνης για τους πολίτες. Και ίσως πρέπει να δούμε ακριβώς και τι δημόσια αγαθά ε, παρέχει ε, το ενίο νόμισμα. Τέλο πάντων, αν θα μπορούσαμε να το δούμε και το ευρώ σε ένα δημόσιο αγαθό. Είπαμε ότι υπάρχει και ο ελέφαντας στο δωμάτιο, δηλαδή οι σχέσεις ευρωζώνης αφενός με τα κράτη που δεν θέλουν να είναι στην ευρωζώνη αφετέρου. Υπήρξαν κάποιοι με το Ηνωμένο Βασίλειο, που δυστυχώς τα έλεγα εγώ, για πρώτη φορά τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης ε, δέχθηκαν την ιδέα ε, μιας πολυνομισματικής ένωσης multi-currency union, αλλά δεν υπάρχει ένα νέο πλαίσιο. Μέχρι στιγμή είμαστε όλοι στο κοινοβούλιο εδώ, κοινοβούλιο της Ευρωζώνης, γιατί όλες οι χώρες είχαν ε, δυνητικά ε, την δυνατότητα να μπουν, λέει το πρωτοκολλο 12, μέχρι να ενταχθούν όλες οι χώρες. Δηλαδή υπήρχε ένα θέμα χρόνου απλά και γι' αυτό και δεν ε, έχουμε δύο διαφορετικά όργανα. Αν όμως επικυρώσουμε αυτή την ιδέα της Πολυνομισματικής Ένωσης, τότε θα χρειάζεται και ένα πλαίσιο. Το πλαίσιο αυτό δεν μπορεί να είναι πια ενιαίο, όπως ήταν μέχρι τώρα, εν αναμονή της προσχώρησης όλων των χωρών στην Ευρωζώνη. Θα κάνω τροπολογίες, φαντάζομαι ότι και άλλοι συνάδελφοι θα συμφωνήσουν μαζί μου. Και κάτι τελευταίο. Υπάρχει ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που σχετίζεται με τους ίδιους πόρους. Ήδη ε, προβληματίζεται από αυτού μια διοργανική ομάδα εργασίας. Ε, το θέμα του ελέγχου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από τα Εθνικά Κοινοβούλια ή από μια μεικτή δομή θα εξαρτηθεί σίγουρα από τις επιλογές που θα γίνουν σε ό,τι αφορά την προέλευση των πόρων. Θεωρώ επειδή πρόκειται για έκθεση πρωτοβουλία, ότι σε αυτό το στάδιο θα πρέπει να κρατήσουμε ανοιχτέ τι επιλογέ και να προσπαθήσουμε να είμαστε αυστηροί. Αν δηλαδή είναι εθνικά τα κονδύλια, θα μπορούσε αυτό να δικαιολογεί η παρέμβαση των Κοινοβουλίων. Αλλά μιλάμε τελικά τότε για προπολογισμό τη Ευρωζώνη ή όχι. Ή θα επαναλάβουμε τις δυσκολίες που έχουμε αντιμετωπίσει μετά τις καταστροφικές αποφάσεις ε, και με την άδεια καρέκλα του Ντεγκόλα το 1966. Μήπως θα ξαναξεκινήσουμε ένα σύστημα ελέγχου ε, όπως γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο λόγω από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Υπάρχει ένα παράδοξο. Ομαδοποιημένα ε, και σωστά νομίζω θέλουμε να ε, ορίζουμε κάποια πράγματα για την Ευρωζώνη. Αλλά και πάλι έχουμε ένα σύστημα που θα ε, κατακαιρματίσει και θα διαχωρίσει όλους αυτούς τους πόρους θέλουμε να διαθέσουμε στην Ευρωζώνη. Είναι καλή βάση εργασία. Θα προβούμε στι τροπολίε να τη βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, όποιο θέλει το λόγο τον έλαβε. Θα ζητήσω τώρα λοιπόν από του δύο συνεισηγητέ να μα πούν ποια είναι τα συμπεράσματά του από αυτήν την πάρα πολύ πλούσια και δημοκρατική συνεδρίαση. Κύριος Μπέγκε. Uh, Πράγματι, κύριε Πρόεδρε, η συζήτηση ήταν ε, πολύ Ε, βεβαίως ε, και υπήρχε και κάποια φυλακτικότητα, αλλά υπήρχε και υποστήριξη που δόθηκε στην εισηγήτρια. Ξεκινάμε με αυτά που είπε ο συνάδελφος Παουλ Τάγκ. Κύριε Πρόεδρε, απαντήσατε εν μέρη και απάντησε επίση και ο κύριος Γκαλτιέρη. Ίσως ε, θα πρέπει όλα αυτά να τα ξαναστείλουμε στους συναδέλφους. Ε, είναι μια έκθεση ε, του 2013 όπου είναι οι νομικές επιλογές για επιπρόσθετη δημοσιονομική ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης του καθηγητή Ρεπάζη. Κοιτάξτε, αυτή είναι μια πάρα πολύ ε, καλή αξιολόγηση με βάση που αυτά μπορούν να γίνουν δημοσιονομικά, το τι επίσης δεν μπορεί να γίνει και το τι μπορούμε να κάνουμε χωρίς ε, ε, συνθηματικές τροποποίησεις. Και εδώ επανέρχομαι σε κάτι που είπε ένας συνάδελφος, δηλαδή υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορούμε να κάνουμε χωρίς τροποποίηση των συνοπτικών, αλλά θα ήταν καλό να επιτύχουμε μια σταθερότερη βάση με συμπληρωματικές διατάξεις. Ε, των συνθήκων. Πράγματι λοιπόν, εδώ ε, συμβαίνει αυτό που είπε ο συνάλφος κύριος Γκουαλτιέρη και όλα αυτά καλύπτονται με την έκθεση που σας ανέφερα. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα στην ιστορία του προεπολογισμού, όπου μπορεί κανείς να ξεκινήσει να δουλεύει με ίδιο πόρους, ε, να σέβεται τους, ε, τα όρια, ίσως και κάποιες φορές ε, να ξεπεράσει τα όρια, παρόλα αυτά ε, να υπάρχουν τα δικαιώματα ελέγχου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έστω και με οποιαδήποτε μορφή. Άρα δηλαδή όλα αυτά είναι εφικτά και ίσως θα πρέπει όλα αυτά να τα διαθέσουμε στους συναδέλφους. Υπάρχουν ε, κάποιες ε, ερμηνείες που ακούσαμε σήμερα ε, για το τι είναι εφικτό και το τι δεν είναι εφικτό. Και θα ήθελα να παρακαλέσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να γίνει λίγο πιο σαφής έτσι ώστε να έχουμε μία επιπρόσθετη βάση συζήτησης. Με βάση όμως την εμπειρία μου στο, στα δημοσιονομικά εδώ και 25 χρόνια θέλω να σας πω ότι όλα αυτά είναι εφικτά κυρίως όταν μιλάμε για εκείνα τα στοιχεία της δημοσιονομικής κανότητας που πρέπει να εισαχθούν συμπληρωματικά. Πρόκειται λοιπόν ε, για το ότι τα κράτη-μέλη θα μπορούν να μεταφέρουν από τον προπλησμό προς τα έξω και το Κοινοβούλιο θα μπορεί επίσης ε, να προβαίνει σε εξωτερική ανάθεση. Όλα αυτά ήδη γίνονται. Άρα δηλαδή όλα αυτά αποδεικνύουν ότι στο πλαίσιο το δημοσιονομικό, των δημοσιονομικών κανονισμών ε, μπορούμε να προχωρήσουμε με αυτόν τον τρόπο. Άρα δηλαδή δεν συμφωνώ με αυτά που είπε ο συνάδελφος από την Ισπανία, από τους ε, σοσιαλδημοκράτες. Μίλησε για δικτατορία των Βρυξελών. Όχι, δεν είναι έτσι. Διαλέξαμε την διακυβέρνηση κυβερνητική μέθοδο και εάν θέλουμε να προβάλλουμε την ενωσιακή μέθοδο, αυτή είναι μια καλύτερη μορφή της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας και της συμμετοχής των κοινοβουλίων. Γιατί έχουμε ε, διπλή, διτή επίδραση και αυτό με ανησυχεί. Ε, υπάρχουν εθνικά κοινοβούλια που και δεν θα συμμετέχουν και δεν θα συμμετέχουμε ούτε εμείς. Άρα δηλαδή στην περίπτωση αυτή έχουμε κοινά συμφέροντα ε, για τα οποία θα πρέπει να συσκεφτούμε και όλα αυτά να τα μεταφέρουμε στα εθνικά κοινοβούλια. Ο κύριος Τάγκα έχει δίκιο ότι όλα αυτά που κάνουμε εδώ δεν επιλύουν τα προβλήματα ούτε και τους ε, προϋπολογισμούς ε, ενός συγκεκριμένου, ούτε ε, τα προβλήματα ενός συγκεκριμένου προϋπολογισμού. Κατηγορίες 3 και 4 νομίζω ότι θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας σε αυτά τα συγκεκριμένα προβλήματα και στο τέλος των, ε, της όλης υπόθεσης ε, φοβάμαι ότι ε, δεν θα μπορούμε να λειτουργήσουμε. Και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Όσον αφορά τη συνάδελφα από τη Φιλανδία, θέλω να της πω ότι το θέμα του moral hazard νομίζω ότι το θίξαμε με απόλυτη σαφήνεια. Και όταν μιλάμε για την ερεσιμότητα και την αλληλεγγύη, νομίζω ότι υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία που έχουν καθοριστεί και όταν αναφερόμαστε σε συναδέλφους σε χώρες που ήδη αντιμετωπίζουν σήμερα το θέμα της ερεσιμότητας, ε, τα κράτη αυτά θα διαμαρτυρηθούν ότι είναι είναι πολύ αυστηρή η αιρεσιμότητα. Σωστό, η αλληλεγγύη και οι προϋποθέσεις ε, είναι άρρηκτα συνδεμένες μεταξύ τους, διότι ε, Πράγματι πρόκειται ε, για επεμβάσεις ε, στα κοινωνικά συστήματα των κρατών μελών και αυτό είναι κάτι που δεν είναι εύκολο. Ε, στο σημείο αυτό θα ήθελα να πω κάτι που έχει σχέση με τις χώρες ευρώ και χώρες εκτός ευρώ. Ε, νομίζω έχουμε πει πολύ προσεκτικά ότι η βασική αρχή είναι η κοινή αγορά και το νόμισμα είναι το ευρώ. Ε, δύο κράτη ζήτησαν εξαίρεση και επτά κράτη κάποια στιγμή πρόκειται να μπουν στο ευρώ. Άρα το μη ευρώ είναι η εξαίρεση σε αυτό το πλαίσιο των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό θέλω να σας δώσω μία συμβουλή. Οι συνάδελφοι οι οποίοι ανήκουν εκτός ευρώ ε, θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί ως προς τις ε, κόκκινες γραμμές ε, να ξέρουν ε, τι είναι απαραίτητο ενδεχομένως για τη σταθεροποίηση της Ευρωζώνης. Το Φεβρουάριο ε, υπήρξε ένα πακέτο, υπήρξαν διαπραγματεύσεις από αυτού σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο και εντάξει μπορεί να μην πολύ αρέσει αλλά τι να κάνουμε. Αυτό όμως είναι το ελάχιστο. Δηλαδή όσοι ε, δεν είναι στο ευρώ, δεν μπορούν να τοποθετούνται επί του ευρώ, ε, γιατί στην περίπτωση αυτή ξεπερνάνε μία κόκκινη γραμμή ε, και όσον αφορά το ενδεχόμενο μελλοντική συνεργασία. Ευχαριστώ τον συνάδελφο Τόμπαλτς και σε παλαιότερε συζητήσει των σκιωδών εισηγητών κατέστησε απόλυτα σαφές το τι ακριβώς σημαίνει το τι ακριβώς θα συνέβαινε αν δεν υπήρχαν τα διαρθρωτικά ταμεία. Όσον αφορά τις προτάσεις που κάνατε, πράγματι αυτή η ομάδα υψηλοπιπέδου για τους ίδιους πόρους θα συνεδριάσει το Σεπτέμβρη και ίσως εκεί μπορούμε να δούμε ε, πώς όλα αυτά θα τα συμπεριλάβουμε στην Ολομέλεια, στην τελική έκθεση της Ολομέλειας. Τα συνταγματικά δικαστήρια έχουν ε, διαπιστώσει ότι υπάρχουν κάποιες δυνατότητες ελιγμών αλλά αυτά σε συνδυασμό με τα εθνικά κοινοβούλια και πρέπει να βρούμε κάποιες λύσεις έτσι ώστε τα προγράμματά μας να μην αποτύχουν. Παρακαλώ κυρία Περέσο έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους κυρίως που μπήκαν στο κόπο να διαβάσουν την έκθεση και συμφωνούν τις προτάσεις. Ο κύριος Μούρεσαν διαστόματος Μπάλτς. Έθεσε ορισμένα ερωτήματα και θα ήθελα να το απαντήσω ότι ο βασικός μας στόχος ως συνεισηγητές είναι να είμαστε συγκεκριμένοι σε κάποια σημεία αφενός, αλλά έχουμε και έναν άλλο βασικό στόχο. Έναν ή δύο μήνες μετά τις ε, διασταφές των σχέσεων ε, με το Ηνωμένο Βασίλειο τον Οκτώβριο να δώσουμε ως κοινοβουλίο ένα σαφές μηνύμα προς τα άλλα θεσμικά όργανα. Αυτό είναι σημαντικό για τη λειτουργία της Ευρωζώνης. Το άρθρο 125 δεν το αναφέραμε γι' αυτό, αλλά διαμακρόν αναφερόμαστε στην ισορροπία των πληρωμών. Και θα δούμε το 125 που εγγράφεται, που εντάσσεται. Σε ό,τι αφορά το αν χρειάζεται αλλαγή της συνθήκης ή όχι με πρώτο τον κύριο Μωρέ, σαν πολλοί συνάδελφοι το ανέφεραν. Πουθενά δεν λέμε ότι δεν θέλουμε αλλαγή τη συνθήκη. Ο κύριο Βάιτσεκερ πολύ σωστά λέει ότι κάποια στιγμή θα χρειαστεί κιόλα να καταγραφεί ότι πρέπει να αναδιατυπωθούν οι δεσμεύσει ε, των κρατών μελών σε σχέση με, το, με τη συμμετοχή του στην Ευρωζώνη. Τι σημαίνει δηλαδή να είναι μια χώρα μέλο τη Ευρωζώνη. δεν μπορούμε να προδικάσουμε, ούτε μπορούμε να παγορεύσουμε ή το αντίθετο ε, να γίνει το οτιδήποτε είναι δυνατό στο πλαίσιο των συνθήκων και ο κ. Γκουαλτιέρη νομίζω πολύ καλά είπε ότι υπήρχε ευελιξία στη συνθήκη. Θα το μελετήσουμε κι εμείς, αλλά μπορούμε να δούμε και να υποβάλουμε προτάσεις που θα μπορούσαν να αποτελούν σημαντικές εγγυήσει για την λειτουργία τη Ευρωζώνη ω Τάνκ επέμεινε στου τρει πυλώνε, την ισορροπία μεταξύ αλληλεγγύη και ευθύνη. Αυτό είναι κάτι που μας βρίσκει σύμφωνος και θέλουμε ε, να είναι ο ηρμός αυτός στην ε, έκθεσή μας. Κυρίως για να αποφύγουμε και την παγίδα ή τέλο πάντων ε, το να μας κατηγορήσουν ότι είμαστε υπέρ ενός ηθικού κινδύνου. Εγώ μάλιστα είμαι από αυτούς που αρνούμε να τα θέσω όλα στο επίπεδο του ηθικού κινδύνου. Γιατί ναι, να το έχουμε υπόψη μας το θέμα αυτό. Το λέμε στην έκθεση, εντάξει, ηθικός κίνδυνος, αλλά να υπάρξει παρόλα αυτά κάποια πρόοδο. Αφού αναγνωρίζουμε όλη τη βροζόνη είναι Σε ό,τι αφορά τώρα την κατανομή των αρμοδιοτήτων, πρέπει να υπάρξουν διευκρινήσει, το είπαν πολλοί. Και αυτό ο κώδικα διοντολογία έχει ω στόχο, συγγνώμη, σύγκληση, έχει ω στόχο την ε, ιδιοποίηση σε εθνικό επίπεδο και τη χρήση εθνικών εργαλείων και την καλύτερη αξιοποίησή του. Ο πρόεδρο Αρτού επανήλθε στη διάκριση μεταξύ προπολογισμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση και προπολογισμού τη Ευρωζώνη. Κατά βάθο τώρα, πώ όλα αυτά θα είναι μετά από 20 χρόνια, τι να σα πω, δεν έχω καμιά ιδέα. Μπορεί να μην υπάρχει πια καμιά διάκριση. Όμω σήμερα βλέπουμε ότι ακριβώ επειδή έχουμε αυτό το νομικό πλαίσιο με 19 κράτη-μέλη στην Ευρωζώνη, 7 που μπορούν δυνητικά να προσχωρήσουν και δύο που έχουν opt-out, πρέπει να οργανωθούμε, πρέπει να οργανώσουμε κάπως αυτή την κατάσταση. Και αυτό κάνουμε με την πρότασή μας. Λέβαια Τόρβαλτς, δεν θα επανέλθω στο θέμα της συνοχής. Α, δεν είναι εδώ ο κύριος Τόρβαλτς, τέλος πάντων. Αυτό ε, λέω για να μείνει στο Δινίκες. Θα του το πούνε και οι βοηθή του. Λοιπόν, γιατί σύγκλησε τα είπε Μπέγκε, για την ιδέα ότι πιο εύκολο είναι το εξάντα από το εξπόστ. Δεν θα στοιχημάτιζα όλες μου τις οικονομίες αυτό, γιατί ήταν πιο εύκολο το εξάντα, τότε μετά το Μάστρ ξέραμε πολύ καλά ότι μπορούσαμε, είχαμε μάλλον κάνουμε ακόμη κάποια πράγματα και αυτό το κοινοβούλιο και στην έκθεση, το είχε πει εκ των εξάντε με την έκθεση μέτων και μετά βιαστήκαμε να μην ασχοληθούμε με θέματα που ήταν στον πυρήνα της λειτουργίας της Ευρωζώνης. Πρέπει να είναι συμπληρωματικές οι δύο προσεγγίσεις. Σίγουρα είναι πιο δύσκολο το πλαίσιο, αλλά νομίζω τώρα πρέπει να τα δούμε αυτά τα ζητήματα. Για τον Μπάσικ Χάουτ ε, συμφωνώ και ευχαριστώ που μας υποστηρίζετε. Στην όλη συζήτηση νομίζω ότι αναδύεται ένα ευρωπαϊκό πνεύμα. Την κίνημα δουλειά φαίνεται αυτό. Για τον ESM, να που κάνουμε μια διευκρίνηση. Πράγματι, ε, στοιχηματίζουμε πολύ σε αυτό το μηχανισμό γιατί έχει μεγάλες δυνατότητες, όμως ε, στις τροπολογίες μας είπαμε ότι θα συμπληρώσουμε την έκθεση μετά από αυτή την ανταλλαγή απόψεων. Νομίζουμε ότι ο ESM θα πρέπει να παραμείνει ως κεντρικό στοιχείο ενός από τα σκέλη δυνατότητας αντίδρασης σε, ασύμετρο σοκ. Αυτό το λέμε ξεκάθαρα στην έκθεση. Δημοσιονομική ικανότητα μεταξύ αυτού του οπλοστασίου είναι και το ESM, αλλά δεν είναι το μόνο όπλο. Και να σας υπενθυμίσω ότι Γι' αυτό το financial backstop λέμε και αυτό ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη στη συζήτηση. Ο κύριος Μαραγκάλ. Μας προτείνει για αυτό το Ταμείο Χαλεπών λοιπόν Καιρών να, κάνουμε, να βάλουμε κάποιες όρους. Κάποιοι όμως ρώτησαν τελικά θα εθετήσουμε έναν αυτόματο μηχανισμό ή όχι. Εμείς θεωρούμε ότι υπάρχουν αιρεσιμότητες, υπάρχουν όροι στο πλαίσιο του ESM όπως λειτουργεί σήμερα. Αν θέλουμε πραγματικό όμως να λύσουμε τα θεωρητικά πρακτικά προβλήματα που έχουν να κάνουν την ύπαρξη της και αντίσταση της Ευρωζώνης στα σύμμετρα σοκ, θα πρέπει να έχουμε νομίζω έναν αυτόματο μηχανισμό. Γι' αυτό και προτείνουμε το Rainy Day Fund Νομίζω ότι έχω απαντήσει σε πολλούς συναδέλφους σε σχέση με αυτό που είπε ο Χάνας Φερνάντες, δύο παρατήσει. Πρώτη, για το EFSM. Στην παράγραφο 22 κάνουμε μία μνήμα σε αυτό το μηχανισμό. Και λέμε ακριβώς ότι σε αυτό το πνεύμα θα πρέπει να το συμπεριλάβουμε σε αυτή την πρόταση για προπολογισμό της Ευρωζώνης και σε ό,τι αφορά τη χρήση των κερδών της έκτα, το είχαμε αναφέρει και στην ακρόαση που έγινε, οι δύο συνεισηγητές συμφώνησαν ότι είναι ένα σημείο το οποίο θα επανέλθει στη συζήτηση με την κατάθεση σχετικών τροπολογιών. Πάρτε στυλό λοιπόν και εμείς θα δούμε Πώ θα τα αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα ζητήματα και το συγκεκριμένο ζήτημα. Και για την τελευταία παρέμβαση τη Σιλβί Γκουλάρ, δημόσια αγαθά κτλ. Σίγουρα είναι κάτι που πρέπει να το σκεφτούμε. Και για την έκθεση του Μάριο Μόντι τώρα, τον οποίο και συναντήσαμε στη Ρώμη, ό,τι καταλαβαίνουμε τελικά αυτή η ομάδα εργασίας αρχικά. Δεν υποτίθεται ότι θα είχε εντολή να ασχοληθεί με το αν θα υπάρχει, θα υπάρχει προπολογισμό ευρωζώνη. Άλλαξε όμω κάπω αυτό. Οπότε μιλά συγκεκριμένα για την Ευρωζώνη. Θα δούμε πώς η ομάδα εργασία ε, θα ε, αντιμετωπίσει και θα χειριστεί αυτό το θέμα και θα δούμε πριν μπορούμε να κάνουμε, αν χρειάζεται να προσαρμόσουμε και την τελική μας διατύπωση περί των Λομέλη. Για να δούμε υπόψη και τη απόψη ομάδας Μόντι. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ την Περβάνς, ευχαριστώ τον Ράιμορ, ευχαριστώ του κοινού συγητές. Σα ευχαριστώ. Πήρατε το λόγο. Θα ήθελα να σας διευκρινίσω ότι η ημερομηνία κατάθεση τροπολογιών προβλέπεται για τις 7 Ιουνίου στις 12. Οι συγητές όμω δεν έχουν πρόβλημα να, καθιστε... να βάλουμε δύο, ώρες αργότερα, ε, δύο μέρες αργότερα, 9 Ιουνίου δηλαδή, 9 Ιουνίου στις 12 το μεσημέρι, η προθεσμία κατάθεσης ε, τροπολογιών. Επόμενη κοινή μας συνεδρίαση Econ Badge είναι, ε, προγραμματισμένη για τις 11 Ιουλίου για να μελετήσουμε τις τροπολογίες αλλά και για να ακούσουμε τους Υπουργούς Οικονομικών που δέχτηκαν να έρθουν να μιλήσουν εδώ στην κοινή μας συνεδρίαση. Πολύ σημαντική στιγμή λοιπόν. Και σίγουρα το Σεπτέμβριο η Επιτροπή μας η ε, Μικτή θα ξανασυνεδριάσει ώστε να αποφασίσει, να ψηφίσει με ε, την προοπτική του, της Ολομέλειας του Οκτωβρίου. Λοιπόν, ροκανίσαμε λίγο χρόνο από την Επιτροπή ΕΚΟΝ. Ζητώ από τον πρόεδρό της να μας συγχωρέσει, αλλά σας βάλαμε και σας μέσα στην παράβασή μας. Ε, εντάξει, εν μέρει είναι και δικό μου το λάθος. Άντε, μόνο 15 λεπτά είναι, νομίζω ότι άξιζε τον κόπο. Ήταν χρήσιμη η σημερινή συζήτηση. Να συγχαρώ και εγώ τους συναδέλφους.